της ημερήσιας διάταξης έχω μια ανακοίνωση. Η κυρία Ιβέτα Γκριγκούλε ε, γίνεται μέλος της ομάδας ΑΛΔΕ με ημερομηνία από σήμερα, 27 Απριλίου και πλέον δεν είναι μια εγγεγραμμένη